Il Presidente. Allora. Care colleghe e cari colleghi, buonasera. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σε όλους. Επαναλαμβάνεται η συνέδρια του Κοινοβουλίου που διακόπηκε στις 22 ε, Νοεμβρίου του 2012. Τα πρακτικά